θα ψηφίσουμε αύριο. Ακολουθούν οι παρεμβάσεις ενός λεπτού και δίνω το λόγο στη, με την κυρία Μποξόρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η, η ειρήνη και η εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι το σημαντικότερο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές χώρες θέλουν να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό συμπεριλαμβάνει και μια σειρά από υποχρεώσεις. Η Ουκρανία αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Ο πληθυσμός της Ουκρανίας έχει και μια ουγγρική μειονότητα 150 και πάνω χιλιάδων ατόμων αλλά η μειονότητα αυτή έχει θίγει από βίαιες ενέργειες εναντίον της, ιδίω η πορεία που έλαβε χώρα το Μάρτιο εφέτος που εστράφει κατά των Ούγγρων. Αυτό στρέφεται κατά του συντάγματος της Ουκρανίας και κατά των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας αυτής. Εγώ υπέβαλα μια γραπτή ερώτηση στην κυρία Μογκερίνη και στην απάντησή της η κυρία Μογκερίνη μου είπε ότι η Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και θα επανέλθει στο θέμα αυτό εάν έχει περισσότερε πληροφορίε. Τσαπάρντα. Το δικαίωμα για την ελεύθερη κυκλοφορία και για την ε, δυνατότητα εργασία οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θεμελιώδε δικαίωμα. Δυστυχώ, πολύ έντιμοι εργαζόμενοι, οι οποίοι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αντιμετωπίσουν διακρίσει εναντίον του. Έχουμε δει πάρα πολλέ περιπτώσει τα τελευταία χρόνια όταν Ρουμάνοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ω πολίτε δεύτερη κατηγορία και αντιμετωπίζουν καταχρήσεις και παραβιάσει σε βάρο του που δεν θα πρέπει να ισχύουν τον 21ο αιώνα. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας, καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει ότι όλες οι ρήτρε των συνδικών σε σχέση με την εργασία την χάνουν σεβασμού. Θα πρέπει να πούμε όχι σε κάθε μορφή διακρίσεων και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση όλων σε σχέση με τα δικαιώματά τους και θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό φορέα για να αντιμετωπίσει τι καταχρήσεις αυτού του είδου στα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι Ρουμάνοι δεν πηγαίνουν στη δύση τη Ευρώπη για να αποκτήσουν χρήματα, αλλά γιατί το τμήμα αυτό τη Ευρώπη του χρειάζεται σε πολλού τομεί. Και έτσι προσθέτουν αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει λόγο που τα λέμε παραβάσει ενό λεπτού. Σα παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε το χρόνο. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Σλοβακία θα είναι η πρώτη φορά που θα αναλάβει τα ενία της Προεδρίας στο επόμενο εξάμεινο και ένα από τα θέματα που θα την αποσχολήσουν είναι η μετανάστευση. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαμε ακούσει δηλώσεις ε, Σλοβάκων πολιτικών για τη μετανάστευση που... Ε, αμφισβητήθηκαν στην Ευρώπη και ε, έκαναν κάποιους να ανησυχήσουν. Ε, πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων και να προστατεύσουμε την Ευρώπη από την τρομοκρατία, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με το καθεστώς των ετούντων άσυλο τα προβλήματα τα οποία ε, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Σλοβακικής Προεδρίας δεν αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ελπίζω να αναλάβει μια πρωτοβουλία και να προσπαθήσει να υπάρξει μια συνένεση που θα διασκεδάσει τις ανησυχίες των, πολιτών και να φροντίσουμε να σεβόμαστε κάθε ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ κύριο Στανασέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Χαιρετίζω την ε, πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών να έχουμε ε, μηδέν ε, περιστατικά HIV-AIDS και περιστατικά υπατήτηδα ε. πρόσφατα έγινε ένα συνέδριο το οποίο ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα. Η φυματίωση είναι η πρώτη αιτία θενάτου για ασθενείς HIV-AIDS. Χωρίς κατάλληλη θεραπεία, 7 στους 10 ασθενείς ε, που πάσχουν από HIV AIDS ε, θα και ε, παθαίνουν φυματίες ή θα πεθάνουν. Πολλοί ασθενείς δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε κατάλληλα φάρμακα. Ε, πρόκειται για περιοχές τις οποίες έχουμε τη μεγαλύτερη μόλυνση από τον ιό HIV AIDS και τα υψηλότερα ποσοστά φυματίωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σχετικό πρόγραμμα εκπνέει φέτος και πιστεύω ότι δεδομένων των συνθηκών θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για το 2016-2020 ώστε να επικεντρωθεί στο HIV AIDS και στη φυματίωση και σε σχετικές άλλες μολυσματικές ασθένειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο αρμόδιος επίτροπος θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται εστονείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσουρκάνου στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στις καταχρήσεις των αρχών προστασίας ε, ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται καταχρήσεις και ε, κακοποίησει σε βάρο οικογενειών Ρουμάνων. Η οικογένεια Μποναβιού είδε πέντε παιδιά να τους ε, παίρνουν από την οικογένειά τους. Πολλέ ε, βέβαια χώρε πίεσαν την Νορβηγία και τελικά θα επανενωθεί η οικογένεια. Το ίδιο έγινε στον Ηνωμένο Βασίλειο με μια άλλη οικογένεια. Δύο εβδομάδες έκανε ο πατέρας απεργία πείνα για να έχει τα παιδιά του. Συνεπώς κάνουμε έκκληση στο Ηνωμένο Βασίλειο για να σέβονται τα δικαιώματα των ανηλίκων και των οικογενειών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάτι για να αποφεύγονται τέτοια δράματα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο βασικό δικαίωμα του ανηλίκου, πρόκειται για τη σύσταση του 89, και την επανένωση των οικογενειών βάσει του άρθρου 9 για τους ανηλίκους. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Καρτον Ντάρλινγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε να πάρουμε μια από τι μεγαλύτερε αποφάσεις για τι επερχόμενε γενιέ στο Ευρωπαϊκό, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το δικαίωμα τη εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θέμα αυτό οι εργατικές ενώσεις ε, εργάζονται και αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ισότητα ανδρών και γυναικών και δυνατότητα εργασίας με ίσες συνθήκες για όλους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα εδραίωσε αυτά το 1982. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει σώσει πάρα πολλές ζωές. Η γονική άδεια, η ίση αντιμετώπιση για ίση εργασία, η ίση μεταχείριση για τους εργαζόμενους σε προσωρινή ή μερική εργασία, το δικαίωμα πληρωμένων διακοπών, όλα αυτά έχουν ε, υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγοντας μια, ένα αγώνα προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή η εκστατεία για την εγκατάλειψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το, από το Βασίλειο δεν αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Ψηφίστε για να μείνει το Ενωμένο Βασίλειο. Παρακαλώ στις 23 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σελίμ Οβίτς έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο χώρες έχουν τη μεγαλύτερη παρουσία σκλαβιά σήμερα, το Ουσβεκιστάν και το Πακιστάν. Είναι δύο χώρες με τις οποίες έχει στενή σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας, μια έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας έδειξε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ηγέτες του Ουσβεκιστάν να συνεχίσουν τις ε, προσπάθειές τους να κρατάνε τα παιδιά στο σχολείο και όχι σαν σκλάβους στην, ε, στο θερισμό του, ε, του βαμβακιού. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι για τα θέματα αυτά και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη έχουν αποστρέψει το βλέμμα τους όταν η καταναγκαστική εργασία των ενηλίκων αλλά και των παιδιών είναι μια μόνιμη πρακτική στι χώρε αυτέ. Η Κομισιόν πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι χώρε αυτέ και να ενισχύσει τον αγώνα κατά τη καταναγκαστική εργασία στην Κεντρική Ασία. Ο Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα το Bundestag ψήφισε καταδικάζοντας ε, κλίματα κατά της ανθρωπότητας ε, στη γενοκτονία των Αρμενίων, όπως γνωρίζετε. Έπρεπε να αποδοθεί ιστορική δικαιοσύνη και αυτό προκάλεσε πολύ περίεργες αντιδράσεις από πλευράς ε, του Τούρκου Πρωθυπουργού. Μία αντίδραση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες και με την πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή και ε, που συγκαλύπτει τα εγκλήματα των τουρκικών αρχών ε, τον καιρό εκείνο. Αυτό το υποστηρίζει και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος. Φοβάμαι λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν πάρα πολλές ε, απαραχωρήσεις σε ένα αυταρχικό καθεστώς όπως είναι το καθεστώς στην Τουρκία. Η κυρία Άντερσον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ριζικέ μεταρρυθμίσει εξού και το ΣΥΝΦΕΝ συμμετέχει επικριτικά. Τα συμφέροντα του Ιρλανδικού λαού δεν εξυπηρετούνται πάντα με τον καλύτερο τρόπο από τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Ούτε και ο βορρά ε, τη Ιρλανδία εξυπηρετείται, οι πολίτε του δηλαδή. Εποφελείται όμως παρόλα αυτά ο Βορράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αγρότες μας, από την κοινή γεωργική πολιτική και τις άμεσες πληρωμές, οι φοιτητέ μας που ταξιδεύουν στην Ευρώπη για να σπουδάσουν και οι επιχειρήσεις μας που έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία αγορά με δυναμικό 500 εκατομμύρια ε, Πελάτε. Μα προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντα εγγύσει για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, για διακοπέ, για ε, δικαιώματα μητρότητα κλπ. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μα προσφέρει η Βρετανική κυβέρνηση. Αν υπάρξει η Brexit, τότε η Βόρεια Ιρλανδία θα είναι δέσμευτη του Ηνωμένου Βασιλείου και απόσχεσταν δεσμευτική. Το Sinn Féin λοιπόν δεν πανηγυρίζει πάντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε εξυπηρετεί πάντα αυτή καλύτερα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολίτων. Παρόλα αυτά, το Sinn θέλει να παραμείνει η, ο βορράς της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Η συνεργατική και η οικονομία ήρθε για να μείνει και πρέπει να υποφεληθούμε από τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή σε μία εναρμονισμένη προσέγγιση στο πνεύμα της εσωτερικής αγοράς και προς το συμφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών οι οποίοι χρησιμοποιούν περισσότερο την ε, ε, κοινή αυτή η οικονομία και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. 36% των καταναλωτών έχουν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή είτε το R&B είτε οτιδήποτε από τα στοιχεία αυτά της συνεργατικής οικονομίας. Και η οικονομία αυτή στην Ευρώπη είναι της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων, έτσι εκτιμάται. Και θα είναι 250 δις την επόμενη δεκαετία από ό,τι φαίνεται. Άρα οι καταναλωτές έτσι έχουν μεγαλύτερη επιλογή, ευελιξία και προσφέρει και ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην οικονομία αυτή δημιουργούν θέσεις απασχόλησης για την τοπική οικονομία. Συνεπώς, χαιρόμαστε για την πρόσφατη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν θέλει ένα πάτσουερ ρυθμίσεων από τις διάφορες χώρες, αλλά αντίθετα υποστηρίζει ένα νέο μοντέλο με προστασία των καταναλωτών, με δίκαια φορολόγηση και αντιμετώπιση των εργασιακών, προβλέποντας πώς θα εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στη συνεργατική αυτή οικονομία. Ευχαριστούμε. Μπέρναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Βόρειο Ανατολική Ακλία έχει πολλά να κερδίσει από την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά να χάσει αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφή τα ωφέλη της παραμονής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή για την απασχόληση, δίνει πρόσβαση στη βορειοανατολική Αγγλία, πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Βοηθάει τις επενδύσεις στις φτωχότερες περιοχές. Παίρνουμε περισσότερα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι δίνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τα δικαιώματα και των εργαζομένων και των καταναλωτών. Μας κρατάει ασφαλή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε τώρα το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι καλή για το αγωτικό τοπίο και το περιβάλλον. Καθαρίζει το νερό μας, προστατεύει τα άγρια ζώα και μας βοηθεί να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή από κοινού. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί και φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μόνος με χώρος που θα βρει κανείς ε, εκτροφή, ε, εκτροφή προβάτων θα είναι μονάχα στα μουσεία. Για μας στην Βορειοανατολική Αγγλία είναι σαφές ότι προτιμούμε να μείνουμε στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Άρκιν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε το συνεχές αυτό πρόσημα ότι για όλα αυτά η Κομισιόν και οι Βρυξέλλες μας έχουν υποχρεώσει να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μην εφαρμόζει κανείς τιμολόγηση του ύδατος εάν δεν το θέλουμε. Το 2010 διευκρινίστηκε ότι μια εδρεωμένη πρακτική θα πρέπει να ισχύει εάν ίσχυε ήδη όταν εγκρίθηκε μια οδηγία. Και αυτό έγινε ήδη από το 2013. Το 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατεδίκασε την Κομισιόν όταν πήγε τη Γερμανία <clears throat> στο δικαστήριο επειδή δεν τιμολογούσε ορισμένες βασικές υπηρεσίες. Το δικαστήριο ήταν σαφές. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αφήνει στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν τα μέτρα που θέλουν για την ανάκτηση κόστους χωρίς να περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την χρήση ύδατος και η οδηγία δεν υποχρεώνει να υπάρχει τιμολόγηση όλων των δραστηριοτήτων για την υδροδότηση. Αυτό που ισχύει για τη Γερμανία πρέπει να ισχύει και για την Ιρλανδία και οι πολιτικοί της Ιρλανδίας που θέλουν να κατηγορήσουν τις Βρυξέλλες το κάνουν για προσωπικό τους κέρδος αλλά δεν έχουν νομική βάση για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σέρπου στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Μία πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι ένα στα τρία παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών είναι είτε υπέρβαρο είτε παχύσαρκο. Το κόστος ε, της θεραπείας των συνοδών ε, νόσων είναι το 1 δέκατο όλων των δαπανών για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά δεν γίνεται καμία ουσιαστική πρόοδος προκειμένου να αναστραφεί αυτή η τάση. Είναι απαράδεκτο η καταπολέμηση της παχυσαρκίας να γίνεται καθαρά στα χαρτιά και να μην υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε καμία περίπτωση. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα διότι πρέπει να έχουν όλοι οτιδήποτε στη διάθεσή τους προκειμένου να αποφύγουν αυτή την απειλή. Ενημέρωσε κατάλληλα τρόφιμα σε κατάλληλες τιμές, προστασία κατά της παραπλανητικής διαφήμισης, ιδίω όταν πρόκειται για προϊόντα για τα παιδιά. Ε, πρόσφατα προτάθηκε πιλωτικό πρόγραμμα για την ε, δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει και εκπαίδευση για την ε, διατροφή. Θεωρώ ότι πρέπει να δίνονται κατάλληλες πληροφορίες και στα παιδιά και στους γονείς και σε νηπιαγωγία για παράδειγμα όταν σχεδιάζουν τα καθημερινά γεύματα των παιδιών. Ελπίζω οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαμίκης στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ εδώ και χιλιάδες χρόνια οι αγροτικές περιοχές παρέχουν τρόφιμα και, άλλες γεωργικές, ε, ε, και άλλους γεωργικούς πόρους. Βέβαια, ε, λόγω της δημογραφικής ανάπτυξης, ε, σύν το χρόνο, με την βιομηχανική επανάσταση, άρχισαν να προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσμο οι πόλες ε, και επομένως ο πληθυσμός των περιοχών της υπαίθρου μειώθηκε. Σήμερα πλέον ο κόσμος ο οποίος ζει σε αυτές τις περιοχές είναι λιγότερος από το 1 δέκατο του συνολικού πληθυσμού και αυτό φυσικά έχει διαφορετικές συνέπειες για την παιδεία, για το κόστος μεταφοράς, για τη στέγαση, διότι υπάρχει μεγάλο κόστος για την πανεγκατάστασή τους όταν φεύγουν από την περιοχή της υπέθρου Επομένως η περιοχή αυτή χάνει την αξία της με κάθε έννοια. Επιπλέον, τα διάφορα κοινωνικά στρώματα ε, είναι σε κίνδυνο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες πλήγονται περισσότερο, ιδίως μετά το 2004. Σας ευχαριστώ πολύ. η κυρία Ρης στη συνέχεια. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μαριάς. Σήμερα, ανήμερα της επαιτίου της απόβασης των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ήττα του ναζισμού, ο Αλβανός Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, σε ένα παραλήρημα εθνικισμού, έθεσε ζήτημα τσαμουριάς, εκπροσωπώντας, όπως είπε, Αλβανούς πολίτες, απογόνους των Τσάμιδων, αυτών δηλαδή που καταδικάστηκαν από την ελλάδα ως εγκληματίες πολέμου μια και ως ένοπλα τμήματα συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της γέρμανο ιταλικής κατοχής με τα ss και τη wehrmacht δολοφονώντας χιλιάδες έλληνες αμάχους. ήρθε λοιπόν η στιγμή η ελλάδα να απαιτήσει πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις και από την αλβανία για τις εγκληματικές πράξεις των τσάμιδων συνεργατών των ναζί ιδίως τώρα που ο πρωθυπουργός της αλβανίας έντι ράμα αναδέχθηκε επισήμω τα δίθεν δικαιώματα άρα και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των τσάμιδων. άλλωστε δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ελλάδα το 1945 δεν αποδέχτηκε τη συμμετοχή της αλβανίας στη διεθνή διάσκεψη ειρήνης των παρισίων μια και η αλβανία όπως άλλωστε και η γερμανία είχε και συνεχίζει να έχει ευθύνες για την αποζημίωση της ελλάδας. τότε η αλβανία αποτελούσε μέρος της ιταλίας του μουσολίνη που επετέθηκε στην ελλάδα το 1945 40 και παρέμεινε μέχρι το 1943 ως δύναμη κατοχής της πατρίδος μου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Next Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τερικάμπρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εχθές, Κυριακή 5 Ιουνίου, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στη Βαρκελόνη υπέρ ε, του ευρώ και τη, του, του πουταμού εύρου και του δέλτα. Η ισπανική κυβέρνηση εξακολουθεί να προτείνει ένα υδρολογικό σχέδιο το οποίο επικρίνουν όλοι οι οργανισμοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί διότι αντιβαίνει στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία ε, λέει ότι δεν θέλει να λάβει αποφάσεις για την κοινωνική πολιτική αλλά και πάλι με το σχέδιο αυτό προσπαθεί να πλήξει τη βιωσιμότητα του Εύρου και του Δέλτα του. Ε, είναι ανεπτές οι οποίες ε, ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να συνεχίσει η βιώσιμότητα ε, και σήμερα θα ήθελα να συμφωνήσω με τους χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούν από την Ισπανική κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο και ζητούν υποστήριξη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμφωνήσει με το αίτημα των πολιτών για να προστατεύσουμε ένα ποταμό ο οποίος είναι ζωτική σημασία για την περιοχή και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Ward. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ, το τάμπινγκ του Χάλιβα από την Κίνα συνεχίζεται στην Ευρώπη με τον Ντέβιτ Κάμερον <clears throat> να είναι ηγέτης μιας μικρής ομάδος ανεύθυνων χωρών που μπλοκάρουν την πρόταση της Κομισιόν για πιο δίκαιους δασμούς που θα σώσουν τη χαλιβουργία μας. Έχω όμως και κάποια καλά νέα. Τα χαλιβουργία στο Βέρμπερτον και στο Σκάρμπορο έχουν αγοραστεί και διατήρησαν έτσι 224 εργασίε στην Κάμπρια που είναι η εκλογική μου περιφέρεια και με τον τρόπο αυτό διατηρούν 4.000 εργασίες στην ε, αλυσίδα τροφοδοσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γαλλία. Οι εργατικοί βουλευτές είναι αυτοί οι οποίοι καταδεικνύουν πάντα την ε, ε, στάση του Κάμερον την ανάλυτη της του Κάμερον έναντι της ε, χαλιβουργία μας. Χάρη στις εργατικές ενώσεις και τον Άλαν Σμιθ έχουμε επιτύχει να σώσουμε τη χαλιβουργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται σε συνεργασία μεταξύ των πολιτικών και των ηγετών της βιομηχανίας και των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, ενιαία αγορά σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και στη δυσλειτουργία αυτής της αγοράς. Στην Ευρώπη έχουμε το δικαίωμα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων που δίνει κάποια υποστήριξη στους πνευματικούς δημιουργούς σε σχέση με τα έργα τους μέσα από τις ε, εταιρείες συλλογής. Αυτό έχει σαν στόχο να κάνει τα έργα προσβάσιμα στους καταναλωτές. Αλλά δυστυχώς έχουν μονάχα οι δημιουργοί τα δικαιώματα μόνο για συγκεκριμένες μορφές καλλιτεχνικών έργων. Δεν υπάρχει συνολική προστασία σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει μια ενιαία αντιμετώπιση. Ευχαριστώ η κυρία Ματίας. Πατήστε το κουμπί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από συστηματικές απειλές προς την Πορτογαλία για κυρώσεις, ε, θεωρήθηκε από την Κομισιόν ότι η Γαλλία δεν πρέπει να υποστεί γιατί η Γαλλία είναι η Γαλλία. Πρέπει οι κανόνε όμω να ισχύουν σε όλους. Ε, για να μπορέσει να υπάρχει σταθερότητα για μερικά κράτη προσπαθεί η Κομισιόν να ε, υποχρεώσει τις χώρες αυτές να κάνουν αυτά τα οποία θέλει ακόμα και αν αυτό οδηγεί σε κατάρρευση της οικονομίας για άλλες σώσεις. Έχουμε μια πραγματική κρίση δημοκρατικής νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια καταστροφή στον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα λόγω της λιτότητας. Μετά από αυτές τις καταστροφές που στις οποίες οδήγησε η πολιτική λιτότητας χωρίς να πετύχει τους στόχους της. Τώρα έρχεται ο της Κομισιόν και λέει ότι τώρα θα σας εφαρμόσω κυρώσεις σε εσά αλλά όχι σε άλλους. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και πρέπει να υπάρξει όχι μόνο αντιμετώπιση οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο νομιμότητας γιατί είναι παράνομα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Κάντε κάτι στην Ευρώπη λοιπόν, τηρήστε τις πραγματικές σας υποχρεώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καν. Κυρία Πρόεδρε, 17 μέρες απομένουν ε, μέχρι το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια απόφαση που δεν θα επηρεάσει μόνο το μέλλον της Βρετανίας, αλλά και κάθε χώρα που είναι εδώ στο Κοινοβούλιο και εκπροσωπείται. Είναι τεράστιες οι συνέπειες. Θα υπάρχει άμεσο οικονομικό σοκ ε, και Τρία εκατομμύρια θέσει εργασία θα είναι σε κίνδυνο. Ε, μπορεί να σταματήσουν να δουλεύουν επιχειρήσει και θα υπάρξουν και συνεργασίε οι οποίε θα κυρωθούν. Η εκστρατεία υπέρ του, ε, της αποχώρησης δεν έχει απαντήσεις. Δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις για την οικονομία και την ασφάλεια και έχουν ε, καταφύγει σε απειλές ε, για τους πρόσφυγες. Τις τελευταίες εβδομάδες λένε ότι όλοι οι μετανάστες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι είτε εγκληματίε είτε ε, δεν έχουν δικαίωμα σε άσυλο. Επειδή και εγώ είμαι μετανάστης, ε, γνωρίζω ότι δεν έχουν καμία βάση αλήθεια σε αυτά τα στοιχεία και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μόνο να προσφέρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και νομίζω ότι οι αξιοπρεπείς άνθρωποι θα το γνωρίζουν και αυτοί και θα υπερψηφίσουν την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στις 23 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Τούμ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η... μιλάω για τους πολίτες που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6% πριν από 24 χρόνια έπαψε να υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολίτες από την Λετωνία και την Εστονία οι οποίοι εξακολουθούν να είναι απάτριδες σύμφωνα με την ε, Ρώσ που είναι απάτριδες στην Εστονία και στην Λετωνία. Έχουν συλλεχθεί υπογραφές με τις οποίες ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι για τους απάτριδες. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Κυρίως για τους Εστονούς και τους Λετωνούς, κυρίως τους Λετονούς, είναι δυσανάλογο το ποσοστό των ανθρώπων αυτών που δεν έχουν δικαιώματα, που είναι απάτριδες. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για τα άτομα αυτά, που είναι απάτριδες στην Εστονία και την Λετωνία. Δεν προβλέπετε μπλε κάρτα στην διαδικασία αυτή. Παρακαλώ, κύριο Φερέρα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος και ο κύριος Δράκη και η παρέα τους κάνουν ας κάνετε μια προσπάθεια να ακούσετε αυτό το οποίο σας λέμε. Ο αγώνας των εργαζομένων και του πορτογαλικού λαού έριξε την κυβέρνηση η οποία ακολούθησε τις κατευθύνσεις σας. Καταδίκασε τις πολιτικές σας ο πορτογαλικός λαός. Ο αγώνας των εργαζομένων και του λαού στην Πορτογαλία ακολούθησε ένα διαφορετικό δρόμο. Αγωνιζόμαστε και καταφέραμε να εξαλείψουμε τις περικοπές στους μισθούς του δημόσιου τομέα και του ελάχιστου μισθού καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την ενίσχυση της, ε, των κοινωνικών παροχών και την προηγούμενη εβδομάδα επανήλθαμε στο ωράριο των 35 ωρών στο δημόσιο τομέα. Όλα αυτά δεν φτάνουν. Θα πετύχουμε πολλά περισσότερα. Κύριε Γιούνκερ, η Γαλλία είναι η Γαλλία, εντάξει, αλλά και η Πορτογαλία είναι η Πορτογαλία μια χώρα με πάνω από 800 χρόνια ιστορίας και με υπερηφάνεια για την ανεξαρτησία της θα χαράξει μόνη της την, ε, τη μοίρα της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γιόνκερ στις 31 Μαΐου πήγε στο συνέδριο των Δημάρχων της Γαλλίας για να τους πει ότι η Ευρώπη είναι αυτή. Όχι κύριε Γιόνκερ, η Ευρώπη είσαστε εσείς. Η πολιτική λιτότητας ε, που έχει κάνει τον κόσμο να πεινάσει είσαστε εσείς. Εσείς είσαστε ο Δήμιος, ο οποίος ε, παριστάνει ότι 27 εκατομμύρια σε 6 χρόνια πήρε η Γαλλία από τα δημοτικά ταμεία, ενώ κοστίζει δύο φορές παραπάνω η Ευρώπη στη Γαλλία για το ίδιο διάστημα. Είσαστε ένα δήμιος που του κοροϊδεύετε όταν τους λέτε ότι η Κομισιόν έχει μια ψυχή, ενώ εσείς εκπροσωπείτε την οικονομική ολιγαρχία που τους ε, πιέζει όσο δεν γίνεται άλλο. Το LuxLeaks, Παναμά ε, κλπ. Όμω ο κόσμο θα καταλαβαίνει όλα αυτά και όλο και περισσότεροι κύριοι Γιούγκερ είναι εκείνοι οι οποίοι σα υπενθυμίζουν ότι εσεί είσαστε ε, ο λακιστή και όχι η εκείνη. Εκείνη αντίθετα είναι οι πατριώτε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαδάκης τώρα έχει το λόγο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλθει στην Ελλάδα αφού καρατόμησε συντάξεις και ασφαλιστικά δικαιώματα παρέδωσε και την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας στα ΦΑΝΣ. Ταυτόχρονα εφαρμόζει άγρια φορολεηλασία εξασφαλίζοντα ζεστό χρήμα για του βιομήχανου και του εφοπλιστές τώρα μάλιστα προετοιμάζει νέο νόμο για τα εργασιακά με όρους γαλέρας αντίστοιχους με αυτούς που περνούν στη γαλλία στο βέλγιο και σε κάθε κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης είναι οι λεγόμενες βέλτιστες πρακτικές της ευρωπαϊκής ένωσης και των οργάνων της όπως το ευρωκοινοβούλιο που βγάζουν τους εργάτες κατά χιλιάδες στον δρόμο. έτσι ακριβώς ονομάζετε εσείς το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού τις ομαδικές απολύσεις τους περιορισμούς στην απεργία όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για την ανάκαμψη του κεφαλαίου είναι ο μαγνήτης για τις επενδύσεις σαν αυτές που μόλις υπέγραψαν οι κυβερνήσεις ελλάδας και γαλλίας στην πλάτη των λαών των δύο χωρών. αποτελεσματική εργατική λαϊκή απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο με τον οργανωμένο ταξικό αγώνα για ανάκτηση των απολειών την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των παρεμβάσεων του ενός λεπτού. Συνεχίζεται αύριο η Ολομέλεια. Θα ξεκινήσουμε στις 9 το πρωί. Έχει ε, δημοσιοποιηθεί η μερίσια διάταξη. Είναι αναρτημένη στο σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρα στη συνεδρίαση.